Λοιπόν, συνάδελφοι, θα αρχίσει η ψηφοφορία. Συνάδελφοι, ευχαριστώ. Θα αρχίσουν οι ψηφοφορίες τώρα, αλλά προηγουμένως την προσοχή σας λίγο σας παρακαλώ. We have a point of order from Madam Hasenkamp. Η κυρία Χάζεκάμπ έχει ένα διαδικαστικό. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κυρία Χάζεκάμπ. Ευχαριστώ πρόεδρε εκατομμύρια ζώων καθημερινά σε όλη την Ευρώπη σφάζονται και θανατώνονται και περιμένουν στα εξωτερικά μας σύνορα. Ένα εκατομμύριο πολιτών ζήτησαν να τερματιστεί αυτή η κατάσταση. 223 μέλη του Κοινοβουλίου ζήτησαν να συσταθεί η Ειδική Εξεταστική Επιτροπή και σήμερα τρία μέλη στην πρώτη σειρά αποφάσισαν ότι δεν το θέλουν. Και τρία, τρία λέξεις έχω να σας πω μόνο στα αγγλικά. Shame on you. Ντροπή σας. Ε, μάλιστα, θα τα διαβιβάσω αυτά τα σχόλιά σας στον πρόεδρο. Ο κύριος Ουρμπάν Κρέσπο. Και εσείς διαδικαστικό έχετε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε. Πρόεδρε. Απόψε δολοφόνησαν τη Μαρια Φράνκο στο Ρίο Ντετζανέιρο, που σύμβουλος του Πεσόλ φεμινίστρια, αντικαπιταλίστρια, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε ένα κλίμα πολιτικής βίας προεκλογικής στη Βραζιλία. Από εδώ θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους συντρόφους και στις συντρόφισσες και να καταδικάσουμε απερίφραστα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το κλίμα βίας που επικρατεί στη Βραζιλία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Ουρμπάν Κρέσπο. Άλλον διαδικαστικό του κυρίου Βιώτη. Did you have a point of order, sir? Διαδικαστικό έχετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να σας ενημερώσω ότι χθε έγινε κάτι το οποίο ήταν ε, τελείως ε, εξωπερίεργος αυτό το μέγαρο. Κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου του κυρίου Σαλβίνη, ο φρουρός τον ακολουθούσε δεν επέτρεψε στον τύπο να του κάνει ερωτήσεις. Δεν επέτρεψε στου δημοσιογράφου να του θέσουν ερωτήσει που όφυλαν να ρωτήσουν και μάλιστα του απείλησαν και σωματικά στο μέγαρο αυτό. Ε, θα πρέπει να επιτρέπετε στου δημοσιογράφου να κάνουν τη δουλειά του. Πρόεδρο. Σα παρακαλώ, συνάδελφοι. Ωραία. Ησυχία, παρακαλώ. Είναι Πέμπτη. Ξέρω ότι θέλετε να ψηφίσουμε και αγωνιάτε. Ανησυχώ πάρα πολύ γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που λέγουν ότι θέλουν να λάβουν το λόγο. Εκτός αν είναι διαδικαστικό, δεν νομίζω ότι μπορώ να το δεχτώ. Η κυρία Μούντι. So I would ask you, please. Σας παρακαλώ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μούντι για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους των συναδέλφων Γκέρλινγκ, Σκοτ Κέιτο και μου της Ιδίας, πρέπει να πω ότι εκπροσωπούμε το Σάλσμπερι από την ε, νότιο-δυτική ε, Αγγλία και πόλη όπου κατοικώ ε, ως υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης βουλευτές πρέπει να πούμε ότι με το ψήφισμα του Brexit για μέσα η εβδομάδα ήταν δύσκολη αλλά κοιτάξτε κυρία Μούντι να σας πω ότι είναι όνειδος αυτό το πράγμα που κάνετε. Κάνει μια δήλωση για ένα σοβαρό θέμα η συνάδελφος. Κυρία Μούντι, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως έλεγα, ως Βρετανή βουλευτή, υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ψήφισμα για τον Brexit περάσαμε δύσκολη εβδομάδα. Έχουμε αμέριστη αλληλεγγύη από το σώμα, από ό,τι είδαμε, στο πλαίσιο όμω επιθέσεων που δεχόμαστε και αυτό το εκτιμήσαμε ιδιαίτερω. Οι ψηφοφόροι μας θα καθησυχάζονται από την ε, βεβαίωση ότι και εσεί θα μα στηρίξετε για να εξασφαλίσουμε ειρήνη και ασφάλεια. Thank you. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μούντι και ακούσατε τα χειροκροτήματα νομίζω. Συγγνώμη κυρία μου, θα σας δώσω το λόγο. Κυρία Άτκινσον, ορίστε, διαδικαστικό ελπίζω να έχετε. μπορώ να ρωτήσω, όχι δεν μπορείτε να ρωτήσετε την κυρία Μούντι για τον ηγέτη του κόμματός της που δεν κατεδίκασε την επίθεση αυτή και εδώ στο κοινοβούλιο. Η Ρωσία φταίει. Συνάδελφοι, δεν είναι ώρα των ερωτήσεων αυτή, ούτε ώρα για συζητήσει και μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στι ψηφοφορίε. Πρώτη ψηφοφορία. Η κατάσταση στι Μαλδίβες.